Are you ready for starting the meeting and then soon starting the voting? Ξεκινήσουμε αγαπητοί συνάδελφοι, κάποτε τη συνεδρίαση. Να ψηφίσουμε και όλες. Α, σιγά σιγά καθίστε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η μερίσια διάταξη εγκρίνεται. Ωραία. Ανακοινώσεις. Ε, διερμηνία σήμερα, όλες οι γλώσσες, εκτός από Μαλτέζικα και Κροατικά. Βουλγαρικά και Φιλανδικά μπορείτε να μιλήσετε μόνο. Δεν θα τα ακούτε. Και κάπου εδώ υπήρχε και ένα τηλεοπτικό συνεργείο. Τα έχει καλέσει, το έχει καλέσει ο κ. Χέτμαν. Θα είναι και στην ψηφοφορία από κατάλαβα. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών. Εγκρίνεται 18 Οκτωβρίου, 5 Νοεμβρίου, 19-20 Νοεμβρίου, 7 Φεβρουαρίου και 19 Φεβρουαρίου. Ενεστώτος. Ωραία. Έκθεση για... Όχι, θα σας πω, με συγχωρείτε, τι έγινε στις ε, τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις. Δυστυχώς ο κύριος ε, Μπάλας ε, Γκίγιομ κολλείεται. Λοιπόν, ο πέμπτος τριμερής διάλογος ήταν πολύ αποτελεσματικός. Όπως και ο τέταρτος γύρος στις 21 Φεβρουαρίου. και οι συζητήσεις εστιάστηκαν στο κεφάλαιο εφαρμοστέα νομοθεσία και συγκεκριμένα στην πρώτερη ειδοποίηση, περίοδο διακοπής, μέγιστη διάρκεια ε, στην οποία κανείς υπάγεται στο κοινωνικό σύστημα του κράτους προέλευσης, διαδικασία αμφισβήτησης εγγράφων, μεταξύ των οποίων και το PDA1, συνέχιση δραστηριοτήτων σε δύο περισσότερα κράτη-μέλη, εφαρμοστεία νομοθεσία για δημοσιογράφους σε ευρωπαϊκά ΜΜΕ και πράξη κατεξοδότηση. Και η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα πότε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων θα σας τα πει ο κύριος ε, Μπαλάς. Ε, ορίστε. Παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη που, που σας ε, διακόπτω, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα ήχου από την γαλλική διερμηνία. Ακούμε μόλις τον ήχο και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, πρόεδρε. D'accord. excusez Το συγγνώμη. Τώρα εντάξει, ωραία. Λοιπόν, όπως έλεγα, ο κύριος Μπάλας ε, κολλείται, αλλά στην επόμενη συνεδρίαση θα σας ενημερώσει για το που βρισκόμαστε στο σημαντικό και περίπλοκο αυτό θέμα. Ωραία λοιπόν, περνάμε στις ε, ψηφοφορίες. Ε, βάλτε τις κάρτες στο μηχανηματάκι. Η ισορροπία εργασιακού και οικογενειακού βίου. Ψηφίζουμε την προσωρινή συμφωνία που προέκυψε από τις δύο οργανικές ε, διαπραγματεύσεις την επιβεβαίωση κορεπέρ στις 6 Φεβρουαρίου. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Και πέρασε. μία ψήφι υπέρ, 3 ε, κατά. Συγχαίρουμε τον εισηγητή για το αποτέλεσμα. Thank you. Ε, then we proceed to ε, the... Σε ευχαριστώ λοιπόν. Περνάμε στην πρόταση σύστασης ε, της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πατήστε τα κουμπάκια. Και πέρασε. 30 υπέρ, 3 ε, ε, κατά 4 αποχές. Thank you, Mr. Σας ευχαριστούμε κύριε Λένερς. Περνάμε στο σχέδιο έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για τον Συντονισμό της Οικονομικής Πολιτικής Πτυχε απασχόλησης και κοινωνικών ζητημάτων στην ετήσια έκθεση του 2019. Ψηφίζουμε την τροπολογία 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρασε. 18 υπέρ, 20 κατά. Καλώς. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 53. Τροπολογία 53. Όχι. Μέρος δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μα εγώ νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να το δούμε. Τροπολογία 53. Και τελείωσε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με μία ψηφοδιαφορά. Θαμ 9 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 57 υπέρ. Κατά αποχές να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρασε. Και δεκτή με 25 ψήφους. Τροπολογία 59 υπέρ κατά, αποχές Συγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές Συγκρίνεται. Τροπολογία 64 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 65 χωριστή ψηφοφορία, μέρος πρώτο υπέρ, κατά, αποχές να επαληθεύσουμε το πρώτο μέρος, άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρασε. Και δεκτή με 22 ψήφους. Μέρος δεύτερο, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 67 υπέρ. Κατά. Αποχές να την ξαναδούμε. Την 67. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρασε. Δεκτή με 20 ψήφους. Τροπολογία 69 υπέρ. Κατά αποχές. Επαληθεύουμε την 69 άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρασε και δεκτή. 22 ψήφοι υπέρ. Περνάμε στην συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εβδομήντα τρία. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Όπως ζήτησε το ΕΛΚ, αλλά το SND έχει ζητήσει ονομαστική ε, ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. 73 το πρώτο τμήμα. πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 26 ψήφους υπέρ. το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. απορρίπτεται με 24 ψήφους κατά. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά η ηλεκτρονική απαλήθευση της 81 άρχεται ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας για την τροπολογία 81. Απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΦΑΜ 14 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 85 κατά τμήματα ψηφοφορία, κατόπιν αιτήματος του ΕΛΚ και ονομαστική κατόπιν αιτήματος των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Το πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. πέρα της ψηφοφορίας. Πρέπει να επαναλάβουμε την ψηφοφορία, διότι υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Τροπολογία 85. Το πρώτο τμήμα. Της 85. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ. Το δεύτερο τμήμα. Επίσης, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 38 ψήφους υπέρ. Το τρίτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία για το τρίτο τμήμα. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 39 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 86. Υπέρ. Ναι, ονομαστική ψηφοφορία έχει ζητήσει το SND. Λήξη της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι, ωραία, και εγκρίνεται με 36 ψήφους υπέρ. ΦΑΜ 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται, καλύτερα όμως να το επαληθεύσουμε. 88 άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με τρεις ψήφους διαφορά. 89 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω πρέπει να επαληθεύσουμε και το αποτέλεσμα της τροπολογίας 89. Ψηφίζουμε ακόμη. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 39 ψήφους κατά. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 93 το πρώτο τμήμα υπέρ. Ονομαστική ψηφοφορία ζητώ, συγγνώμη λέει η Πρόεδρος. Λήξη της ψηφοφορίας. Με 22 ψήφους υπέρ εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, επίσης ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 38 ψήφους υπέρ. Συμβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση της συμβαστικής 19. Αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 21 ψήφους υπέρ. ΦΑΜ 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά ηλεκτρονική επαλήθευση της 103. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας για την 103. απορρίπτεται με διαφορά δύο ψήφων. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΦΑΜ 16 το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΦΑΜ 1 Κατά τμήματα ψηφοφορία, το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση, για να είμαστε βέβαιοι. Το δεύτερο τμήμα της ΦΑΜ 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 32 ψήφους υπέρ. ΦΑΜ 2. Κατά τμήματα ψηφοφορία, το πρώτο τμήμα υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση, δεν είμαι βέβαιη. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 25 ψήφους υπέρ. ΦΑΜ 2 το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. ΦΑΜ 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ΦΑΜ 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ΦΑΜ 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΦΑΜ 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΦΑΜ 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 113. Ονομαστική ψηφοφορία. Κατόπιν ετοίματος του S&D. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 21 ψήφους υπέρ. 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση της 116. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας για την 116. Εγκρίνεται με 20 ψήφους υπέρ, 117 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση της 118. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 20 ψήφους κατά. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση της 119. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται με 20 ψήφους κατά 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. 120. Αρχή της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας. Ζητώ συγγνώμη, εγκρίνεται με 25 ψήφους υπέρ. ΦΑΜ 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ΦΑΜ 8 δεν την ψηφίζουμε. 121 υπέρ. Κατά. Δεν τολμώ να πω ότι απορρίφθηκε ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Λήξη της ψηφοφορίας για την 121. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 122 υπέρ. Κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση 122. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. απορρίπτεται με 27 ψήφους κατά. 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές αναφορές 1α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά 7α μαζί με την 8β είναι πανομοιότυπες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Αιτιολογική αναφορά 8α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8γ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε σε αιτιολογικές σκέψεις. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση της 17. Αρχή της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 25 ψήφους κατά. Τροπολογία 18. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ, κατά, αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας 19, αρχή της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας, εγκρίνεται με διαφορά 6 ψήφων. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας 23. Αρχίζει η ψηφοφορία, λήξη της ψηφοφορίας, απορρίπτεται με διαφορά τεσσάρων ψήφων. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση της 31. Άρχιζει η ψηφοφορία, λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με τρεις ψήφους διαφορά. Φαμ G. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τριάντα έξι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Φαμ άλφα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Φαμ ε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Φαμ Δ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Φαμ F κατά τμήματα ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά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 Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε με 31 ψήφους υπέρ και 6 ψήφους κατά. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον εισηγητή. This one now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 για την θέσπιση μέτρων εκτακτού ανάγκης ε, ή στο πλαίσιο του συντονισμού των ε, συστημάτων κοινωνική πρόνοια μετά την απόσταση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να είμαστε έτοιμοι εφόσον αυτό συμβεί. Συμβαστική 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, καταπίπτουν όλες οι άλλες. Και επομένως ψηφίζουμε επί του τροποποιημένου σχεδίου ονομαστική ψήφος παρακαλώ ψηφίστε. Πέρασε. 36 υπέρ, μία κατά. Σας ευχαριστώ. Those Όποιος δεν τρέχει να προλάβει την επόμενη συνεδρίαση, καλείται να παραμείνει ώστε να ακούσει την κυρία Σούκοβα αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Απασχόληση γνωστή και ως ΕΜΠΛ. η οποία θα μας ε, κάνει μια παρουσίαση για τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Νομίζω ότι ήσασταν εδώ πολύ πρόσφατα. Τώρα βεβαίως ελάβαμε αποφάσεις που σας επιτρέπουν να είστε ακόμη πιο συγκεκριμένοι. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Ήμουν πριν από ένα μήνα εδώ. Παρουσίασα την έκτη τροποποίηση του κατεξιότησης κανονισμού. Διακόπτη η Πρόεδρος. Παρακαλώ να μην έχουμε πηγαδάκια την ώρα που ακούμε την εκπρόσωπο της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Έλεγα ότι πριν από ένα μήνα παρουσίασαν την έκτη του κατεξιότητας κανονισμού για, τη, για τις απλωστημένες επιλογές σχετικά με τη χρηματοδότηση του ΕΚΤ στα κράτη-μέλη. Έβδομη τώρα τροποποίηση. Και μέχρι εδώ έχουμε καταφέρει να διαχειριστούμε και να εγκρίνουμε όλες τις προτάσεις των κρατών μελών συμπεριλαμβανομένων των επιλογών απλουστευμένου κόστους που αποστέλλονται, υποβάλλονται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα κράτη-μέλη. Η παρουσίασή μου θα είναι στην κανονική της δομή, λέει η ομιλήτρια. Υπό το άρθρο 14.1 εξιωτείται η Κομισιόν ώστε να υιοθετήσει απλουστευμένες διαδικασίες κόστους σε σχέση με οποιαδήποτε δράση και που μπορούν να υποβληθούν από οποιοδήποτε κράτος μέλος ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι επιλογές αυτές μπορεί να είναι κατά ή κόστος μονάδος και υπό τον κανονισμό τα κράτη-μέλη εκτιμούν ιδιαίτερα την δυνατότητα αυτή διότι τους παρέχεται σαφήνεια δικαίου σχετικά με τις δαπάνες που υποβάλλονται. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιούν εθνικές λογιστικές πρακτικές για τη σχέση μεταξύ δικαιούχων και αρχής διαχείρισης όπως παρέχει και ο κανονισμός κοινών διατάξεων που διέπει τη σχέση μεταξύ Κομισιών και Αρχής Διαχείρισης. Για οποιαδήποτε λοιπόν δράση ή και κάποια επιχείρηση που εμπίπτει στις προϋποθέσεις εθνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες προμήθειες και εκεί μπορούν να επιλέγονται αυτές οι διαδικασίες σε απλουσταμένου κόστους. Υπάρχει ισχυρή πολιτική δεσμευσή και η Κομισιόν διατηρεί το επίπεδο της ασφαλείας της αφιλοδοξίας της να επιτύχουμε το 50% του ESF του ΕΚΤ μέσω απλουστευμένων διαδικασιών για όλα τα κράτη-μέλη που θέλουν οι δικέ του εθνικέ τέτοιε διαδικασίε, διευθετήσει να έχουν εγκριθεί και θα πάμε σε 7 κράτη-μέλη πιο συγκεκριμένα αργότερα. Ο κανονισμό είναι σχετικά περιορισμένο, 4 άρθρα, αλλά επικαιροποιούμε τα παραρτήματα, ένα για κάθε κράτο μέλο Έχουμε ορισμούς για τους δείκτες ε, της ε, μονάδης μέτρησης και όταν τα κράτη-μέλη έχουν παρέχει τα σχετικά στοιχεία μπορούν να επαναδιαπραγματευτούν το κόστος μονάδος επί τη βάση νέων οικονομικών στοιχείων. Μέχρι στιγμής είχαμε έξι λοιπόν όπως έλεγα τροπολογίες για τον κανονισμό που ε, ενεκρίθηκε το 2015 και καλύπτουν 19 κρατημέλη. Αυτό δεν είχε αλλάξει, ο αριθμός δηλαδή των κρατών μελών. Και η Κομισιόν έχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη δυνατότητα να υιοθετήσει απλουσταμένες διευθυντής κόστους, χωρίς περαιτέρω ανάλυση ή δικαιολόγηση. Μέχρι στιγμής τέσσερις τέτοιες διευθυντήσεις έχουν ε, επιλεγεί σε ενωσιακό επίπεδο για τις ε, δημόσιες υπηρεσίες, την κατάρτιση των, των υπαλλήλων. Οι τελευταίες τρεις ήταν μέρος της έκτης ακριβώς τροπολογίας. η οποία χάρη και στην Επιτροπή σας ε, θα τεθεί ενισχύ μέσα Μαρτίου. Η έβδομη τροπολογία που τώρα υποβάλλουμε προς την προσοχή σας τροποποιεί για Γαλλία, Τσεχία, Μάλτα, Ιταλία, Ολλανδία, Κροατία και Ηνωμένο Βασίλειο τα παραρτημένα. Αναχώρα, μπορώ να σας πω, ότι η 7η τροπολογία δίνει νέο κόστος μονάδας για την Ρινιό για προγράμματα κατάρτισης και βασίζεται στο αποτέλεσμα η Κομισιόν θα καταβάλει για κάθε συμμετέχοντα που θα έχει λάβει τίτλο που θα εγκρίνει επίσημη αναγνωσμένη επαγγελματική ένωση, σύλλογος, και για δεξιότητες και κατάρτιση που έχει ληφθεί υπό την συγκεκριμένη επαγγελματική εξειδίκευση. Για την Τσεχία. Λάβαμε μια πρόταση και αντιστοίχω επικαιροποιήσαμε για πέντε μονάδε κόστου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μα επιβλήθησαν θα ήθελα να σα πω ότι η Τσεχία είναι υπαριθμόν ένα στη χρησιμοποίηση τέτοιων διευθετήσεων απλουσταμένου κόστου. Έχουν ήδη 32 τέτοιε. Για τη Μάλτα. Νέα πρόταση για καταποκοπήν ποσά στην περίπτωση έμμεσων δαπανών. Επομένως θα καταβάλλεται κατά κοπήν εφόσον μάλλον στην περίπτωση πραγματικού και άμεσου κόστους δαπάνης. Αυτό επί τη βάση του είδους δικαιούχου και της κλίμακας της επιχείρησης για την Ιταλία έχουμε νέο κόστος μονάδος για την κατάρτιση σε τεχνικό Ινστιτούτο, αντίστοιχο ΤΕΙ e δηλαδή, και σύμφωνα και με τις ώρες κατάρτισης που έχουν συμπληρωθεί ένα έτος. Επίσης, σε σχέση με προγράμματα κινητικότητας για ερευνητές, υπό το πρόγραμμα έρευνα και κοινοτομία. Η Ολλανδία Ωραίο κόστο μονάδα για, την, για τις θέσεις απασχόλησης σχετικά με ανθρώπου με αναπηρία και στην Κροατία νέο κόστο μονάδα για άλλες ε, ευάλωτε κοινωνικέ μονάδες για το Ηνωμένο Βασίλειο που προφανώς το αντιμετωπίζουμε ω κράτος μέλο, λέει ο Μιλήτρια ε, τέσσερα μάλλον νέα, νέες μονάδες κόστους Μιλούμε για ωραίο κόστος για μερικώς απασχολούμενων και ετήσιο ποσοστό το οποίο διαιρείται ανά μήνα. Αυτά, εν πάση είναι τα επτά κρατημέλη και οι διάφορες ε, δράσεις υπό τις διαφθετήσεις από τους κόστος με χαρά να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να έχετε. Βεβαίως, λέει η Πρόεδρος μπορούμε να ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε την κυρία Σούκοβα. Agnes, you look like you want to put η Άγνες μου μοιάζει ότι κάτι θέλει να ρωτήσει, λέει η πρόεδρος. Όχι, λέει η Άγνες. Έχουμε κάποια ερώτηση για την κυρία Σούκοβα. Όχι. Είναι πολύ το σαφή όλα αυτά που μας είπατε, κυρία Σούκοβα. Τώρα το χρονοδιάγραμμα, λέει η Πρόεδρος, έχει ω εξή. Προθεσμία υποβολής οποιασδήποτε αντίρρησης είναι 15 Μαρτίου. Και προθεσμία για το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συνολικά για αντιρρήσει είναι 15 Απριλίου. Επομένως, εάν καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει κάτι προς το οποίο έχετε αντίρρηση, υπάρχει ακόμη ένα περιθώριο, με τελική προθεσμία τέτοιων παρατηρήσεων και αντιρρήσεων από Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, όπως είπα, 15 Απριλίου. Για τις επόμενες συνεδριάσεις δεν έχουμε ακόμα επιβεβαιωμένες ημερομηνίε, θα, το λάβει, θα τις λάβετε το των δυνατών. Έχουμε πολλά ακόμα που πρέπει να χειριστούμε στην Επιτροπή Πρωτού ολοκληρώσουμε την εντολή, τη θητεία και ελπίζω ότι θα έχουμε αποτελέσματα των τριμερών διαλόγων που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα ως τότε να έχετε μια όμορφη βραδιά. Σας ευχαριστώ.